Τα μέλη της Επιτροπής ε, Αναπτύξεως παρακαλώ να καθίσουν πάλι. Να συνεχίσουμε με το υπαριθμό 14 που είναι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. με εισηγήτρια την κυρία Ζόφκο. Ρωτώ την κυρία Ζόφκο, θέλετε να πείτε τίποτα πριν από την ψηφοφορία. Ζελιάνα, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καθώς επίσης ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην σύνταξη της εκθέσεως δεν είχαμε κανένα μεγάλο θέμα. Μου φαίνεται ότι η πρόταση είναι καλή. Θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να βελτιώσει στο μέλλον την πολιτική προστασία και τώρα μάλιστα που έρχεται και η θερινή περίοδος και να μην λησμονούμε ότι πέρσι διακόπτει η Μα πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Σας παρακαλώ εκεί πίσω στην αίθουσα. Αν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ έξω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι η Ένωση αντιμετώπισε βαριές τραγωδίες. Θυμάστε τις ε, πυρκαγιές στην Πορτογαλία, Κροατία και Ιταλία. Με την πρότασή μας ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουμε στην βελτίωση του συστήματος πολιτικής προστασίας και ελπίζω οι συνάδελφοί μου να με υποστηρίξουν στην προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ. Έχει γίνει πρόταση, λέει η Πρόεδρος. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Υπάρχει ένσταση. Διότι έχουν θετικό πρόσημο όλες οι, ε, όλα τα τμήματα της ψηφοφορίας. Όλες μαζί λοιπόν, παρακαλώ ψήφι υπέρ των τροπολογιών. Κατά. Όχι, νομίζω δεν είστε κατά, έτσι είναι. Ε, είστε υπέρ, έτσι είναι. Ναι, ναι. Κατά, λοιπόν, τώρα. Αποχές εγκρίνονται ομόφωνα. Και ονομαστική για την τροποποιημένη πλέον πρόταση. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, καμία κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Ζόφκο. Ακολουθεί ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση για την συμφωνία μετά την Κοτονού. Είμαι η συγκίτρια εγώ ίδια. Δέστε αν έχετε τη λίστα ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, να επαληθεύσω την 2, εντάξει. Τροπολογία 2 λοιπόν. Ξεκολουθεί να ψηφίσετε τροπολογία 2. Τώρα ψηφίσατε όλοι όσοι επιθυμείτε. Ωραία. Τέλος. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. 11-11. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τροπολογία 3 αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι όσοι επιθυμείτε. Ωραία. Τέλος. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση και εδώ. 4. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Όπως τροποποιήθηκε τώρα, συνολικά δηλαδή, η προφορική ερώτηση αρχίζει, εννοείται την ονομαστική ψηφοφόρια, τέλος, εγκρίνεται ψήφι 21 υπέρ, μία κατά. Ευχαριστώ πολύ. Η προφορική ερώτηση θα υποβληθεί δεόντως. Έχουμε τώρα και το ψήφισμα για την προφορική ερώτηση για το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση εδώ 30 επαλήθευση αρχίζει ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 κατά τμήματα πρώτο τμήμα της 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 36. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. 38 υπέρ. Ε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Επαλήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε. 43 επαλήθευση αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται πάλι 11-11. Έγινε η ψηφοφορία τώρα αγαπητέ κύριε Ντέβα. 42. Δεν μπορείτε να διορθώσετε ψηφοφορία μετά από το κλείσιμο ούτε στην Ολομέλεια ούτε και εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να διορθώσετε ψηφοφορία αυτή στην Ολομέλεια πλέον. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ναι αυτή εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 σε δύο τμήματα αυτή πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 σε τρία τμήματα εδώ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Πρώτο τμήμα 54, αρχίζει. Τέλος, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, επαλήθευση. Τρίτο τμήμα της 54, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να επαληθεύσουμε. 55 αρχίζει η επαλήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα, κατά τμήματα 56, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά επαλήθεση 59 αρχίζει νομίζω ότι απορρίπτεται τέλος απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά επαλήθευση αρχίζει πέρας εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, α αυτή καταπίπτει. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70, 75 έχει καταπέσει. Όχι, λέτε όχι. Mm. Α, α, συγγνώμη, λάθος. Επιστρέφουμε στην 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79, 79 υπέρ, κατά. Συγγνώμη λέει η Λίντα, 77 77. Υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση της 77. Επαλήθευση λοιπόν 77 αρχίζει. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Κλείνει τώρα. Μάλιστα, απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση, επαλήθευση. 79. Αρχίζει. Ψηφίσατε. 79. Πέρας. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση 81. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, οι εισηγητικέ σκέψει 6 υπέρ Τροπολογία 6. Να το ξαναδούμε. Επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Να ξαναδούμε λοιπόν. Επαλήθευση της 7 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές. Ίδια πλειοψηφία, άρα εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 12 αρχίζει Πέρας. νομίζω ότι εγκρίνεται και όντως εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να επαληθεύσουμε. Αρχίζει. Τέλος. Απερίφθη. 14. Όλες μαζί. 14, 15, 16. Είστε λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ έτσι είναι 18 λέει τώρα η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όλες μαζί τώρα για τα citations. 1 έως 5 προς το τέλος. 1 έως 4. 1 έως 4 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του σχέδιου ψηφίσματος ονομαστικά. Ανοίγει, πέρας, 21 ψήφοι υπέρ, ούτε μία κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Έχουμε και άλλες όμως ψηφοφορίες. Πρόκειται για την έκθεση, μάλλον είναι σχέδιο γνωμοδότησης για την παραβίαση δικαιωμάτων ηθαγενών σε, ανά τον κόσμο μεταξύ αυτών των παραβιάσεων και αρπαγές γεών με εισηγήτητα την ίδια Χόιμπουχ. Έχουμε λοιπόν συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβολογία, ε, Συμβαστική Β υπερκατάποχε εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπερκατάποχε εγκρίνεται. Γ δηλαδή. Τροπολογία 8 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά επαλήθευση εδώ. Επαλήθευση δεύτερο τμήμα τη 8. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα δούμε. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό. Συμβαστική όχι. Απλώς τροπολογία. Τροπολογία 11. Υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι την 11 τέλος εγκρίνεται συμβαστική D, δέλτα υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται επαλήθευση συμβαστική D νομίζω ότι εγκρίνεται αρχίζει τέλος Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές 22. Ας επαληθεύσουμε λέει η πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Γιατί το μείον είναι σε παρένθεση. Α, καλά, καλά. Ωραία, λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία για την 24. Υπάρχουν στάσεις. Ψηφίζουμε τότε την 24. Την προφορική μάλλον. Υπέρ, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση για την 35. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Α, είχατε δίκιο. Απερίφθη. 37 επτά υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 37 αρχίζει τέλος εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική έτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 45. Ε, Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I, Ι, υπέρ κατά αποχές, επαλήθευση. Συμβαστική I, Ι. Ψηφίσατε, πέρας, πέρας λέω, εγκρίνεται 12-10. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 και 61 καταπίπτουν. Έρχεται η συμβαστική κάπα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές, επαλήθευση, επαλήθευση για την 63. αρχίσει. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά. Επαλήθευση της 65 αρχίζει. πέρα εγκρίνεται. Συμβαστική L λάμδα υπέρ κατά εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 69 αρχίζει ψηφίσατε τέλος απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 τώρα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση πέρας απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας 11-11 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ Α, επαλήθευση για την 77, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας λέω. Εγκρίνεται. 81 τελευταία ε, τροπολογία ψηφίζεται, υπέρ κατά εγκρίνεται. Στο σύνολο του τώρα το κείμενο, με ονομαστική ψηφοφορία, έχει αρχίσει. πέρας 14 υπέρ καμία κατά και 8 αποχές σας ευχαριστώ όλους και όλους πολύ ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Χόιμπουχ Τώρα ακολουθεί το 17 το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας. Η εισηγήτρια λέγεται Μαρία Νόιχλ. Είναι παρούσα. Δεν έχει τίποτε να πει κάποιος πριν αρχίσουμε. Πρόκειται για γνωμοδότηση που γίνεται για λογαριασμό της Επιτροπής Γεωργίας. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 21. Ψήφι υπέρ, δεύτερο τμήμα της 21. Ε, το βλέπετε στο, στη λίστα ψηφοφορίας στην ε, παράγραφο 3α νέο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση της 22 ε, αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι διαμορφώνει την ίδια πλειοψηφία. Χωρίς να είμαι σίγουρη. Ψηφίσατε. Πέρας εγκρίνεται. 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση. Πρώτο τμήμα της 24. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 12-10. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. απορρίπτεται αυτό. 25 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 6. Συμβαστική 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινεται. Ακολουθεί η τροπολογία 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί η 45. Αλλά μόνο το δεύτερο μέρος, το δεύτερο τμήμα της. Υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση, επαλήθευση. Γιατί δεύτερο τμήμα της 45. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Αρχίζει. 50, 50, όχι 60. 50, 5, 0. Ψηφίσατε. Πέρας. περίφθη με ισοψηφία. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μια στιγμή θα κάνουμε παλήθευση, επαλήθευση για την 60. Πέρας. Εγκρίνεται. Σωστό λοιπόν που επαληθεύσαμε. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά. Επαλήθευση για την 63. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά. Επαλήθευση, επαλήθευση 66. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. Ωραία. Τώρα, η γνωμοδότηση του σύνολό όπως τροποποιήθηκε, με ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 15, 0, 7. 15 υπέρ, 0 αποχές και μάλλον 0 κατά και 7 αποχές. Τώρα, ακολουθεί κοινή συνεδρίαση. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, η πρόεδρος. Μια στιγμή. Να ευχαριστήσουμε τον Νικολά, ο οποίος αποχωρεί από την Επιτροπή μας και πηγαίνει στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων και μετά θα πάει στην Ουάσιγκτον, στο γραφείο ε, που εκπροσωπείται εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλή σου τύχη, Νικολάη. Και ίσως να τον δείτε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή και στην Ουάσιγκτον. Τώρα, θα γίνει κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΙΝΤΕ. Έχουμε και πέντε προσκεκλημένους